παίρνετε για να μπορούμε να συμμετέχουμε και να έχουμε παρουσία σε, στο πλαίσιο διεθνών ε, ομάδων. Φυσικά το κοινό σχέδιο υλοποίησης είναι το βασικό μας εργαλείο. Εμείς ε, είμαστε επιφορτισμένοι με την υλοποίηση ακριβώς αυτού του κοινού σχεδίου. Τώρα όσον αφορά πιο συγκεκριμένα την υλοποίηση των ελέγχων για τις εκφορτώσεις και τη μη απόρριψη των παραλιευμάτων. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη. Έχουμε παρουσία στη σχετική ομάδα και θα διοργανώσουμε ένα σεμινάριο για τα κράτη-μέλη όπου θα στείλουμε κάποια βασικά μηνύματα. Σίγουρα χρειάζεται και σε επίπεδο δηλώσεων να κάνουμε κάτι περισσότερο σχετικά αφορά τις απορρίψει εν ώψη της εφαρμογής των κανόνων του 2015. Έχουμε καταρχήν τις δηλώσεις δηλαδή τι απορρίψει που πρέπει να γίνουν εν του 2015 και μετά θα βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη με βάση καλέ πρακτικές να συμμορφωθούν ακόμη περισσότερο με τις υποχρεώσει εκφόρτωσης. Θα δούμε με τα κρατη τι είδους διατάξεις πρέπει να περιέχει ένα πρόγραμμα απορρίψεων το οποίο δεν θα δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση που δεν θα μπορεί να ελέγξει κανείς. Όσον αφορά την ανάπτυξη δυνατοτήτων, η υπηρεσία μας θα συνεχίσει φυσικά μεταξύ άλλων να δουλεύει πάνω στην πληροφορική βασική σημασία για να μπορέσει η υπηρεσία να αντεπεξέλθει στη μείωση του προσωπικού και να βελτιώσει βεβαίω και την διαλειτουργικότητα μεταξύ των κρατών μελών. Ο κανονισμός προβλέπει ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών και το οποίο θα οδηγήσει σε οικονομίε κλίμακα και θα βελτιώσει και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Ως τώρα αντιμετωπίσαμε εμπόδια στον τομέα αυτών, τα οποία επιλύουμε με την βελτίωση της πληροφορικής. Μετά δουλεύουμε πάνω στο σύστημα Fishnet. Είναι το σύστημα το οποίο ενοποιούμε διάφορες λειτουργίες. Δεξάγουμε τηλεδιασκέψεις. Έχουμε ένα σύστημα ανταλλαγής ε, email και στοιχείων με τρόπο αυτοματοποιημένο. Αναφέρουμε τις εκφορτώσεις, απορρίψεις, VMS. Ε, Πρόκειται για μια πλατφόρμα επικοινωνίας λοιπόν που διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επικοινωνία αλλά και την κατάρτιση και την ανάπτυξη των σχετικών ε, προγραμμάτων κατάρτισης. Σε εργασία με τρίτες χώρες. Και εδώ όλο και καλύτερα και πάλι όμως εξαρτώμεθα από την απόφαση, την έγκριση της Κομισιόν. Δεν μπορούμε να πάρουμε δηλαδή πρωτοβουλία χωρίς την έγκριση της Κομισιόν. Είμαστε σε επαφή με τις χώρες του Βορείου Ατλαντικού όσον αφορά τα πλαγικά είδη και τα άλλα είδη της ζώνης ΝΑΦΟ στην Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Συνεχίζουμε επίσης να έχουμε επαφές με τα υποψηφία κράτη και με τις τρίτες χώρες. Το 2014, κατά πάσα πιθανότητα, η Κομισιόν θα ζητήσει από την υπηρεσία μας να διεξαγάγει σεμινάρια κατάρτισης και να λάβει τη δημιουργία ικανοτήτων σε αφρικανικές χώρες κατά το οποίο βεβαίως θα πράξουμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και του προπολογισμού. Μια άλλη δυνατότητα, λιγότερο, λιγότερο πιθανή, αφορά τον κανονισμό για την αδηλωτή αναρχή και παράνομη αλία. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα πώς θα κάνουμε περισσότερα με λιγότερα όπως λέμε. Δουλεύουμε με ενθουσιασμό, όμως ε, φοβούμαι ότι θα χρειαστεί να επικεντρωθούμε στους βασικούς μας ρόλους, τον επιχειρησιακό συντονισμό και την ανάπτυξη δυνατοτήτων. Σήμερα ήδη συνεργαζόμαστε βεβαίως στο πλαίσιο ενός ε, χαρτί πορείες με διάφορους οργανισμούς και αρχές ευρωπαϊκούς και άλλους θα προσθεθούν και άλλες συνεργασίες. Παρά την μείωση του προσωπικού. Χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο νέες τεχνολογίες, από τις οποίες βεβαίως εξαρτώμεθα, αλλά θα είμαστε πιο ευέλικτοι εκεί που τα πράγματα ήδη έχουν προχωρήσει. Εκχωρούμε δηλαδή δυνατότητες ε, συντονισμού αν θέλετε και ασχολούμαστε περισσότερο με τις περιοχές που πραγματικά του χρειάζονται. Εμείς δεν χρηματοδοτούμεθα από τον κεντρικό προπολισμό όπως ίσως ε, γνωρίζετε. Παρ' όλα αυτά είμαστε επιφορτισμένοι με πολλούς ρόλους και καθήκοντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε τη δημιουργία μιας ομάδας η οποία θα εξετάσει την κατάσταση των διαφόρων υπηρεσιών, εξωτερικών υπηρεσιών της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ρεσία έγινε και διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε ότι ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών μας έχει προστιθεμένη αξία. Ε, αυτό έγινε από εξωτερικό αξιολογητή. Επίσης εκφράστηκαν ε, θετικά σχόλια για την υπηρεσία μας όσον αφορά την κανονικότητα και την νομιμότητα των δεπανών μας μεταξύ άλλων όπως προείπε το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθεί να συγκεράσει τις διάφορες τάσεις που εκφράζονται στο δημοσιονομικό πεδίο. όπω είπα, εγκρίθηκε ομοφόνος μια δήλωση προς Κοινοβουλίο, Συμβούλιο, Κομισιόν. Το θέμα για μας από εδώ και πέρα είναι να μοιραστούμε τη δουλειά, να συνεργαστούμε με οργανισμου όπως η ΕΜΣΑ, για την επιτήρηση στη θάλασσα και ούτω καθεξής. Θα ήθελα Εν κατακλείδη να πω ότι η αποστολή μας είναι απαραίτητη, είναι υψηλού επίπεδου, αφορά το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία, υποστηρίζει την αηφορικότητα και την ίδια την ευρωπαϊκή αλία. Δεν υπάρχει αηφορία χωρίς ελέγχους. Δεν είναι μόνο διαχείριση των ικανοτήτων. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες αηφορίας της ευρωπαϊκής αλίας. 20% των αποθεμάτων βρίσκονται στα ωριά τους αυτή τη στιγμή. 39% το 2015 θα είναι αυτά τα αποθέματα. Ο ρόλος πλέον, ο κύριος ρόλος διαδραματίζεται από τα κρατή μέλη. Οι πόροι πηγαίνουν στα κράτη μέλη για να ελοπίσουν ακριβώς αυτές τις ε, υποστηρικτικές δραστηριότητε. Η υπηρεσία μα βεβαίω παραμένει το κέντρο το οποίο φροντίζει την ομοιομορφή εφαρμογή αυτών των κανόνων. Προσπαθούμε και εμείς να συμβάλλουμε στην υλοποίηση της νέας αλληλευτικής πολιτικής. Η υπηρεσία μας θα επιτρέψει μεταξύ άλλων στα κρατη να κάνουν οικονομίες κλίμακας. Παρά το μικρό μας μέγεθος, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής Πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε στους ενδιαφερμένους τα μέσα και τις ικανότητες. Παρά το γεγονό ε, τη μείωση του 1% το οποίο αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τι δραστηριότητέ μα. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, όπως πάντα, θα αρχίσουμε με έναν γύρο ερωταπαντήσεων. Ο αντιπρόεδρο Στίβενσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σαουρέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Πάντα στηρίζαμε τις εργασίες της υπηρεσίας σας. Θα χάσετε έξι μέλη του προσωπικού σας, τη στιγμή που την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσαμε την αναθεώρηση τη μεταρρύθμιση στην κοινή αλλιευτική πολιτική, την οργάνωση των αγορών. Αυτό λοιπόν θα δημιουργήσει πολλές νέες υποχρεώσεις για την υπηρεσία σας. Περιφερειοποίηση, απορρίψεις. Διασφάλιση της ε, μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για τα εμπορικά είδη. Ακόμα και με την αφοσίωσή σας που αναφέρατε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα κάνετε περισσότερα με λιγότερα. Αναρωτιέμαι γιατί τα κράτη-μέλη συχνά στα δικαστήρια τους, εάν κατηγορούνται αλληλείς για παράνομες εκφορτώσεις ηχθείων, Μερικές φορές τα πρόστιμα είναι τεράστια. Στη Βρετανία μπορεί να μιλάμε για εκατομμύρια λιρών. Λόγω της ανάγκης των κρατών μελών να συμμορφώνονται με την πολιτική περιφερειοποίηση δεν υπάρχει δυνατότητα τα πρόστιμα αυτά να διαβιβάζονται στην υπηρεσία σας διότι σίγουρα εάν η αύξηση του προϋπολογισμού σας είναι λιγότερη από, την, από τον πληθωρισμό, θα χρειαστείτε περισσότερα χρήματα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους χρηματοδότησης της υπηρεσίας σας και ίσως τα κράτη-μέλη να μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ. Είναι η δεύτερη φορά που έχω την ευκαιρία να σας ακούσω. Εσείς ε, μιλάτε για την έλλειψη των πόρων και διαμαρτύρεστε γι' αυτό. Έλλειψη πόρων ώστε να ε, μπορέσετε να διαχειριστείτε τις, ε, την, την, ε, τον οργανισμό σας και δεν αμφιβάλλω γι' αυτό ε, αλλά εμείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο μπορούμε να θέσουμε ερωτήσεις στη διάρκεια της εξέτασης του προϋπολογισμού και τέθη μια ερώτηση τον Μάρτιο σχετικά ε, σε εσά την υποβάλαμε, αλλά δεν λάβαμε απάντηση. Οι ε, αρμοδιότητες σας είναι βρύτατες και κατά συνέπεια θα πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί ε, συνεργασίας ώστε να υπάρχει επαρκής έλεγχος της αλίας. Από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν ε, διστάχμοι ανάμεσα σε, στους διάφορους που συνεργάζονται, ενώ αλλού όχι. Όμως το θέμα του ελέγχου, το οποίο θα πρέπει να αναλάβει η ίδια Μήπως θα πρέπει να γίνει πιο επιτακτικό, ε, ίσως να μην θέλετε να μου απαντήσετε εδώ για το ποιοι δεν συνεργάζονται. Πάντως θέλω να έχω μια απάντηση. Και υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι υπάρχει τέτοια ε, έλλειψη ελέγχου. Ποιος επαληθεύει πώς ε, γίνονται οι πληρωμές σωστά, δηλαδή ε, πρέπει να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί κάνουμε πολύ φασαρία, αλλά τελικά στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Και ο κύριος Στίβενσον έκανε μια πρόταση, πολύ καλή κατά τη γνώμη μου, η χώρα μου έχει κάνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση κατά της παράνομης αλληλείας, με τεράστια φορολογική απάτη για τον τόνο, ένα σκάνδαλο αποκαλύφθηκε. Βέβαια υπάρχουν ε, νομικές πτυχές που θα πρέπει να μελετηθούν, αλλά ίσως και ένα τμήμα των ε, οικονομικών κυρώσεων, του πρόστιμου που θα επιβληθεί, θα μπορούσε να δοθεί στον οργανισμό. Υπάρχει ωστόσο κάτι το οποίο με ανησυχεί, γιατί νομίζω πως δεν μπορεί να είναι ε, μόνο ένας χώρος ε, ή οργανισμός που θα κάνει ελέγχους εάν δεν συμπληρώνεται και από τους απαραίτητους πόρους ώστε να ε, προβεί τους ελέγχους που οφείλει. Πώς θα λειτουργήσει αν δεν έχει τους απαραίτητους πόρους. Και είναι αλήθεια πως αυτή η πολιτική λιτότητας και περικοπών που γίνονται τελείως αδιακρίτως δεν βοηθάει. Θα ήταν σημαντικό λοιπόν να δοθούν περισσότεροι πόροι στον ελεγκτικό μηχανισμό που καταπολεμά την υπεραλίευση και την παράνομη αλία. Είναι ουσιαστικό να υπάρχουν και να σας δοθούν περισσότεροι πόροι. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Είναι όπως στο σπίτι μας, στο νοικοκυριό. Δεν θα πανούν όλα τα ίδια πράγματα, εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι η εξή. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ε, τα τελευταία χρόνια μειώθηκαν οι πόροι σας. Οι πόροι δηλαδή τόσο η οικονομική όσο και η ανθρώπινη. Και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πέρυσι κάναμε μια αλλαγή, μια τροπολογία. Ε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Και τελευταία μου ερώτηση. Πιστεύετε πως ε, είναι παθητική η στάση, ότι ο κόσμος δηλαδή δεν συνεργάζεται παραμένει έτσι απαθής. Γιατί εφόσον δεν υπάρχει συνεργασία από την πλευρά των κρατών μελών, είναι δύσκολο και ο οργανισμός να είναι ε, αποτελεσματικός. Ιδιαίτερα στην καταπολέμηση αυτού του προβλήματος ε, με τον ερθρό ή άλλα είδη. Τα ψάρια δεν στέκονται σε μια θέση και οι λαθροαλείς ούτε και αυτοί. Αυτά είχα να πω και κλείνω την παρέμβασή μου. Η αντιπροσωπεία μου και η ομάδα μου σας στηρίζουν. Εγώ η Δία σας υποστηρίζω και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου ώστε να πληθύνουν οι πόροι και να μπορέσετε να ασχίσετε πραγματικό έλεγχο. Θα πρέπει να δούμε βέβαια και ποια ήταν η εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Να δούμε γιατί δεν υπάρχει στα γραπτοκείμενα. Ευχαριστώ κυρία Ρόντου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με την άποψη ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Έχουμε τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Ε, πρέπει να κινήσουμε πολλά πράγματα εντός των κρατών μελών. Την σχετική συζήτηση την είχαμε πριν κάποιους μήνες. Δεν επιτρέπεται τέτοια περικοπή του προϋπολογισμού. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο παράλογο είναι να περικόπτεται ο προϋπολογισμός και να επιβάλλονται νέες υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την υπηρεσία και ό,τι μπορεί να κάνει η πολιτική μου ομάδα θα το κάνουμε. Διότι έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, το έχουμε πει αυτό σαφώς και άλλες φορές. Έχουμε τώρα κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες χώρες χρησιμοποιούν την κατάρτιση που προσφέρεται για τους ε, ελεγκτές. Αυτό το κάνουν ε, όλα τα κράτη-μέλη ή μόνο κάποια. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω τα σεμινάρια που οργανώνεται στα κράτη-μέλη ή που προσφέρεται στα κράτη-μέλη πραγματοποιούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη ή υπάρχει συγκεκριμένη πελατεία που συμμετέχει. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές ερωτήσεις μου. Και εσείς τι μας προτείνετε. Κατά τη διάρκεια της νέας θητείας θα πρέπει να υποβληθεί νέος κανονισμός περί ελέγχου, ποια πράγματα θα πρέπει να προσέξουμε, ώστε ήδη το 2014 να μπορέσουν να λειτουργήσουν έτσι οι έλεγχοι, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί η νέα κοινή αλληλευτική πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ρόδουστ. Η κυρία Λεβέν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σαβουρέ που ήρθατε εδώ και μας παρουσιάσατε την δουλειά που κάνετε. Μας παρουσιάσατε και τις προσδοκίες από την υπηρεσία στο μέλλον, μετά την υιοθέτηση της νέας κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμά αντιλαμβάνονται ότι αυτή θα οδηγήσει σε περισσότερα καθήκοντα για την υπηρεσία σας και περισσότερες προσδοκίες από πλευράς των Ευρωπαίων πολιτών. Ζητούν να ανταποκριθούμε σε αυτά που έχουμε θεσπίσει στο νέο κανονισμό και φαντάζομαι ότι περιμένουν από εμά να μπορούμε να ελέγξουμε αυτά που συμφωνήσαμε. Να μην είναι δηλαδή απλά κενά λόγια σε χαρτί, αλλά να υπάρξει και σωστός έλεγχος των μέτρων. Καταλαβαίνω ότι η υπηρεσία σας ε, πλήττεται από αυτές τις περικοπές του προϋπολογισμού. Τη στιγμή που έχετε και νέα καθήκοντα. Η ερώτησή μου είναι αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται οι διαπραγματεύσεις για τον νέο Ταμείο Αλίας και Θάλασσας. Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιείται τριμερής διάλογος. Το Κοινοβούλιο αύξησε τα ποσά για τον έλεγχο και την συλλογή δεδομένων στη δική μας θέση για το Ταμείο. Κατά 100% μάλιστα έχουμε αυξήσει τα νούμερα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, υπάρχει κάποιος τρόπος ε, με τα χρήματα αυτά να στηρίξουμε την υπηρεσία σας. μπορούμε να σας στηρίξουμε έμεσα μέσω των κρατών μελών ή υπάρχει τρόπος για την Κομισιόν και την ίδια την υπηρεσία να ζητήσει περισσότερα χρήματα. Βέβαια, αυτό εναπόκειται και στα κράτη-μέλη και τα επιχειρησιακά προγράμματα, αλλά σίγουρα πολλά κράτη-μέλη εποφελούνται από την υπηρεσία με τα κοινά προγράμματα κινητοποίησης. Και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, πολλά κράτη-μέλη αλλιεύουν εκτός της Ευρώπης και αναφέρατε ότι η Κομισιόν σας ζήτησε να εκπαιδεύσετε επιθεωρητές στη Δυτική Αφρική. Κάτι το οποίο σίγουρα συνάδει με αυτά που χρειαζόμαστε. Πρέπει να διασφαλίσουμε να είναι βιώσιμη και η εξωτερική διάσταση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει προστιθέμενη αξία και για τις χώρες εταίρους μας. Τα κράτη-μέλη λοιπόν που ενδιαφέρονται για βιώσιμες συμφωνίες αλληλείας με άλλες χώρες θα πρέπει να συνεισφέρουν κιόλα. Και όλοι έχουμε σημαντικές προσδοκίες από την εφαρμογή του κανονισμού για την καταπολέμηση της ε, παράνομης λαθρείας και άναρχης αλληλείας. Έχει ζητηθεί και από εσά να συνεισφέρετε. Είναι τεράστιο το έργο να ταξιδεύει κανείς σε όλον τον κόσμο και να δει πώς τα διάφορα κράτη-μέλη πληρούν ή όχι τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αναγνωριστούν ως εξαγωγής ηχθείων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας περιμένουν λοιπόν σημαντικές προκλήσεις και καθήκοντα. Αναφερθήκατε στην περιφερειοποίηση, αναφερθήκατε και στην Επιτροπή Συμμόρφωσης. Αυτό ήταν μια ιδέα του Κοινοβουλίου, να δημιουργηθεί μια νέα Επιτροπή Συμμόρφωσης. Εσείς την ονομάζετε Ομάδα Εργασίας, άσχετα από το όνομα όμως. Θα πρέπει αυτή η ομάδα, η Επιτροπή, να αποτελέσει ένα εργαλείο για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση από τα κράτη-μέλη με την απαγόρευση απορρίψεων, ώστε να μην είναι ένα μέτρο αυτό το οποίο θα μείνει μόνο στο χαρτί. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 7 δισεκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Γνωρίζουμε ήδη ότι δεν έχουν απορροφηθεί όλοι οι πόροι. Θα μπορούσαν λοιπόν να χρησιμοποιηθούν για την υπηρεσία σας. Αυτή είναι μια ιδέα που ήθελα να αναφέρω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Νομίζω όμως ότι αξίζει τον κόπο να εξερευνήσουμε την ιδέα αυτή περαιτέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Λεβέν. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που να ζητάει το λόγο. Ξαναδίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Σαβουρέ για να απαντήσει στις, απαντήσεις, για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις, ε, στις οποίες θα απαντήσω με τα χαράς. Καταρχήν ε, για τον κύριο Στίβενσον να πω πως πιστεύω πως όντως οι συνομοθέτες εν τη σοφία τους προέβλεψαν τη δυνατότητα στο νέο κανονισμό, το βασικό κανονισμό για την ε, κοινή αλληλευτική πολιτική. Προέβλεψαν λοιπόν να ζητήσουν τον αλληλευτικό τομέα να χρηματοδοτήσει ένα κομμάτι των δαπανών για τον έλεγχο. Ε, εδώ υπάρχει ίσως μια δυνατότητα, ίσως μέσω των κυρώσεων των διοικητικών ή των ποινικών, ανάλογα με την εσωτερική οργάνωση κάθε κράτους μέλους, υπάρχει σίγουρα κάποια δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διάταξη του κανονισμού. Επιπλέον, ε, ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα μέσα στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού κανονισμού να ε, χέρει του side revenue, δηλαδή εσόδων που συλλέγονται μέσα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, όπως είπατε κύριε Στίβενσον, ή μέσω ενδεχομένως ορισμένων πιστώσεων του Ευρωπαϊκού ε, Ταμείου ε, Αλίας, όπως το υπογράμμισε η κυρία Λόβιν. Ε, όσον αφορά τη γραπτή ερώτηση, σας ε, ζητώ συγγνώμη κυρία Γκαρσία Καρβάλια, γιατί σας απάντησα, αλλά σας απάντησα μέσω της διαδικασίας και δεν, με εκπλήσει που δεν πήρατε ποτέ την απάντηση. Σας διαβεβαιώ πάντως πώς θα σας απαντήσω γραπτός. Ε, για τα κράτη-μέλη, να πω ότι η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη είναι καλή. Αλλά βέβαια μιλάμε για το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να ενεργήσει ο οργανισμός μας, ε, το οποίο έχει προκαθορίσει η Κομισιόν. Νομίζω λοιπόν πως οι σχέσεις είναι καρποφόρες, ε, η συνεργασία υπάρχει και κυρίως χάρη στο πρόγραμμα του, της κοινή ε, ανάπτυξης έχουμε, εδώ και έξι χρόνια έχουμε βελτιώσει πολύ την αποδοτικότητα των ελέγχων στην Αλία. Αντίθετα, η ανάπτυξη του συστήματος πληροφορικής εκεί προκλήθηκαν δισταγμοί γιατί αυτό το σύστημα δίνει μεγαλύτερη διαφάνεια και είναι προφανές ότι ορισμένα κρατή-μέλη ανησυχούν για την ε, κοινοποίηση ορισμένων στοιχείων και το θέμα της διαφάνειας είναι ένα θέμα ε, πολύ λεπτό. Εγώ θεωρώ πως είναι πολύ θετικό ε, στοιχείο γιατί έτσι μπορεί κανείς να δει τι ακριβώς κάνει και να μπορέσει να ενεργήσει για να βελτιώσει την επιχειρησιακή του εικόνα, ώστε να είναι πιο σύμμορφη με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί και που έχουν προβλεφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπηρεσία, ο οργανισμός μας δεν έχει κατασταλτική ε, εξουσία. οι ε, δυνατότητες ε, δράσεις ε, ανήκουν μόνο στα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε εμείς να παρέμβουμε. Όμως γνωρίζουμε τις παραβάσεις που γίνονται και έχουμε αναπτύξει μια ομάδα εργασία έτσι ώστε οι αποδείξεις να ε, συλλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι ευρωπαϊκές δικαστικές αρχές στα κρατημέλη που είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους να έχουν αποδείξεις για την παράβαση χωρίς να υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης τη διαδικασία για τυπικού λόγους. Τώρα, όσον αφορά τη δημοσιονομική εξέλιξη, ο προπολογισμό έχει επανέλθει στη βάση του 2012. χωρίς την παρέμβαση έκτακτων πιστώσεων που είχε αναφέρει το Κοινοβούλιο για να μπορέσουν να γίνουν καλύτερα οι έλεγχοι, να ενταθούν οι έλεγχοι. Σήμερα λοιπόν ο οργανισμός σε μια βάση που ήταν αυτή του 11 και του 12 και που θα είναι και η ίδια για το 2013 και 2014 με μια διαφορά 250 ευρώ είναι λοιπόν μια βάση που είναι παγωμένη στην ουσία με κάποιες αναπροσαρμογές που θα συνδεθούν με τον πληθωρισμό. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα κατάρτισης, εμείς διοργανώνουμε κατάρτιση στο σύνολο των κρατών μελών τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή ε, θέλουμε να αναπτύξουμε ε, κατάρτιση στο πλαίσιο της κοινή ανάπτυξης δυνάμεων, ας πούμε για τον ερυθρό τόνο στη Μάλτα ή στην Ιταλία, όπου ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να στείλουν όλους τους επιθεωρητές που κινητοποιούνται κατά τη διάρκεια της επόμενης περίοδου του τόνου ε, και έχουμε κάνει σημαντικές προσπάθειες ε, και στην προετοιμασία της Κροατίας για την είσοδο στην Ένωση. Έχουμε ε, αναπτύξει τρία μαθήματα, το ένα για το IUU το άλλο για γενικά θέματα της πολιτικής αλληλείας και πρέπει να πω πως τα πράγματα πήγαν εξαιρετικά καλά και ότι η ενσωμάτωση της Κροατίας ιδιαίτερα για την περίοδο του Ερθρουτώνου πήγε πάρα πολύ καλά και ήδη έχουμε έναν Κροάτι ελεγκτή στην επιχειρησιακή μας ομάδα Τώρα το θέμα της υποδοχής από, από τις χώρες δεν τίθεται αυτό το θέμα γιατί ο οργανισμός είναι αυτός ο οποίος ε, χρηματοδοτεί το σύνολο των ε, καταρτήσεων, ε, χρηματοδοτεί και τα διπορικά είναι τώρα θέμα του κράτους μέλους αν θα δεχτεί ή όχι την κατάρτιση γιατί ούτως ή άλλως τα οικονομικά, το οικονομικό σκέλος καλύπτεται από τον οργανισμό. Τώρα, τι θα πρέπει να προσέξουμε τώρα για το μέλλον. Το θέμα της, ε, των δυνατοτήτων σε σχέση με τον πόρο. Δηλαδή, δυνατότητες ε, αλίευσης, όπως λέει η ICAT, αυτός ο προβληματισμός είναι ενδιαφέρον και έχει γίνει για τα θυναλιευτικά κυρίως, ε, γιατί σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση όχι μόνο ελέγχου, αλλά έλεγχο που συνδέεται με τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του πόρου. Για μένα είναι επίσης σημαντική η διαφάνεια, δηλαδή η κινητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων φορέων είτε είναι ε, διοικητικός μηχανισμός, είτε είναι οι επαγγελματίε του κλάδου, η κοινωνία των πολιτών, όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίε έτσι ώστε η διαφάνεια και η γνώση για αυτόν τον πόρο που δεν είναι ιδιοκτησία μιας ομάδας ατόμων αλλά είναι ιδιοκτησία του συνόλου των συμπολιτών μας και άρα πρέπει να ε, γίνονται όλα αυτά μέσα στη διαφάνεια και θα πρέπει να έχουν όλα αυτά ε, τη θέση τους στον νέο κανονισμό που προβλέπεται. Τώρα, ένα νομικό θέμα. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και το οργανισμός του Βίγο για τον έλεγχο της δεν ε, είναι επιλέξιμος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλασσίων ε, Υποθέσεων. Δεν έχουμε δυνατότητες πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια παρά μόνο μέσω προγραμμάτων που μπορεί να κάνουν τα κράτη-μέλη, δηλαδή υπό τη μορφή επιχειρησιακών ε, δαπανών, κάποιο προσωπικό που μπορεί δηλαδή να συγχρηματοδοτηθεί από τα κράτη-μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Αλληλεία ή ίσως αν υπάρχουν συνόδοι, συνεδριάσεις, αποστολές, κατά που ε, συγχρηματοδοτείται από τον οργανισμό ή και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας ώστε να γίνουν οικονομίες κλίμακας μέσω δηλαδή του κράτους μέλους πάντα. Το θέμα των συμφωνιών ε, εταιρικής σχέσης ε, για την Λία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για το μέλλον. Ε, Βάλλονται κονδύλια. Τώρα βέβαια το θέμα είναι αν οι εν λόγω χώρες θα δεχτούν να χρησιμοποιήσουν ένα τμήμα αυτών των κονδυλίων για να ε, πληρώσουν το κόστος κατάρτισης ε, στον οργανισμό. Είναι ένα θέμα λεπτό που θα πρέπει να συζητηθεί και όσον αφορά την Επιτροπή Συμμόρφωσης εκεί η υπηρεσία, ο οργανισμός μας είναι παρατηρητής, είμαστε όμως κινητοποιημένοι και ξέρετε ότι αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή ένα σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Ελπίζω πως αυτό το μοντέλο που θα υπάρξει στο τέλη του 2000, θα, θα υλοποιηθεί στο τέλη του Ιουλίου, Ιουνίου 2014 θα μπορέσει όντως να αξιολογήσει αυτά τα θέματα με επιστημονικό και αμερόληπτο ε, τρόπο. Voilà, je pense que répondu... Αυτά νομίζω πως απάντησα και αν κάτι ξέχασα σας παρακαλώ να με συγχωρήσετε εκ των προτέρων. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποια παραπάνω ερώτηση, κάποια ακόμη ερώτηση. Όχι. Ωραία λοιπόν, ολοκληρώνεται εδώ αυτή η συνάντηση και... Α, κυρία Ρόντουστ. Θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε πιο συγκεκριμένα στην ερώτησή μου Ποιες χώρες εποφελούνται από τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Δεν μου απαντήσατε. Ενδιαφέρονται εξίσου όλα τα κράτη-μέλη. Ή υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες εποφελούνται μόνο αυτές και συνεχώς από τις καταρτήσεις των ελεγκτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να ακούσουμε ταυτόχρονα δύο ερωτήσεις και μετά να απαντήσει ο κύριος Σαβουρέ. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ξέχασα να αναφέρω ότι η Ιζαμπέλ Τομάς είναι άρρωστη, θα συμφωνούσε όμως ε, απολύτως με την έκθεση που έχετε συντάξει. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Σαβουρέ. Λυπάμαι, δεν ήμουν ίσως αρκετά σαφής. Η οργάνωση των κοινών ε, σχεδίων σημαίνει ότι όλα τα κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν, ας πούμε στην Βορειοθάλασσα, καλούνται σε σεμινάρια κατάρτισης. Στον Ιάνφο ή στη Βαλτική ή οπουδήποτε αλλού. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων συμμετέχει το 100% των εμπλεκομένων κρατών μελών. Η Ελλάδα δυστυχώς που αντιμετωπίζει δυσκολίες δεν συμμετείχε σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν έχει συμμετάσχει αρκετά, ούτε καν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά είναι μια εξαίρεση η οποία επιβεβαιώνει τον κανόνα. Και ούτως ή άλλως ε, αυτό συνδέεται με την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση στην εν λόγω χώρα. Επίσης, δηλώνασαμε κατάρτιση για τις ε, περικλειστές χώρες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για την Αρχή Παρνάμι Αλία. Πήγαμε στη Βιέννη για να ενημερώσουμε τους ε, επιθεωρητές με αφορμή τη στην Ουγγαρία, την Τσεχία, την Αυστρία βεβαίως και Είχαμε επίση και αιτήματα από συγκεκριμένα κράτη-μέλη να τα βοηθήσουμε για την παροχή κατάρτιση σε εθνικό επίπεδο. Δεν συμβαίνει πολύ συχνά αυτό, αλλά χάρη στη διαθεσιμότητα του νέου προγράμματος κατάρτισης για επιθεωρητές, είναι ένα πρόγραμμα για τις ε, εκφορτώσεις είναι έτοιμο σε 15 μέρες και χάρη και σε άλλα προγράμματα κατάρτισης παράνομες εκφορτώσεις κλπ. Ε, όλο και περισσότερο κράτη-μέλη θα ζητούν τη βοήθειά μας κάθε φορά που θα διοργανώνουν δηλαδή κάποια σεμινάρια κατάρτισης. Τα αιτήματα είναι περισσότερα από χώρες που έχουν εθνικά προγράμματα κατάρτιση. Ε, Κροατία, Γαλλία, Ιταλία. Στον Ηνωμένο Βασίλειο επίση ε, οργανώνουμε κάτι τον Οκτώβριο για θέματα αντίλου τη παρανομή Η κυρία Τωμά ε, είναι υπεύθυνη για αυτά τα προγράμματα. Πολύ ωραία, είχαμε το σημείο 10 της μέρη της διάταξης. Απαλλαγή 2012, για την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελεγχολίας. Πρόκειται για έκθεση επιτροπής προπολογισμού, Το περασμένο καλοκαίρι η υπηρεσία δημοσίευσε την ετήσια έκθεση της, τον ετήσιο απολογισμό, με ε, Το ελληνικό συνεδριό ενέκρινε και η Επιτροπή μας αποφάσισε ο πρόεδρος να συνθέσει την σχετική έκθεση. Την έχετε λάβει νομίζω να πω δύο λόγια όμως περιληπτικά. Εν με την έκθεση αναγνωρίζουμε τη σημασία του έργου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Πιστεύουμε με βάση τα κριτηριά μας ότι διεκπαιρεώθηκαν εκπαιδεύτηκε η εντολή τη με τον σωστό τρόπο. Η υπηρεσία δραματίζει έναν όλο ένα σημαντικότερο ρόλο στο πλαίσιο της νέας ελευτικής πολιτικής στον τομέα της επιτήρησης, της παρακολούθησης και των ελέγχων. Διασφαλίζει έτσι καλύτερο συντονισμό για την επίτευξη των στόχων της, κοινωνικής, της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Εντείνονται οι επιθεωρήσεις αν και καταγράφω την ανησυχία του Διευθυντή, είναι βέβαιο ότι περισσότερους ελέγχους με λιγότερα χρήματα δεν μπορούμε να έχουμε. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου Αλίας να πρικοδοτηθεί με τους απαραίτητους πόρους για να μπορέσει να συνεχίσει να διεκπαιρεώνει ελέγχους όπως έκανε ως σήμερα. Για του ελέγχου χρειάζεται προσωπικό. Είναι απλό. Κατά τα άλλα δεν έχω κάτι άλλο ιδιαίτερο να επισημάνω. Οι ελεγκτέ υπογραμμίζουν την κανονικότητα και νομιμότητα των δαπανών. Το ελεγκτικό συνέδριο επίση συνεχάρει την υπηρεσία για την εξαιρετική, εξαιρετικά αποτελεσματική χρήση των πιστώσεων υποχρεώσεων και πληρωμών. Έχει σημασία όσο μικρό και να είναι ένα προπολογισμό να βλέπουμε ότι όντω οι πιστώσει αξιοποιούνται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Και η έκθεση καταλήγει επισημένοντα τις προσπάθειε βελτίωση των διαδικασιών εντό τη υπηρεσίας και δι όσον αφορά τι δημόσιε συμβάσει και τις προμήθειες. με λοιπόν να χορηγηθεί η απαλλαγή στον διευθυντή Τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου Αλλιές για τον προπολογισμό του 2012. Όλα αυτά περιλαμβάνονται και στο σχέδιο έκθεσης που συνέταξα εκ μέρους της Επιτροπής μας. Αν έχετε ερωτήσεις προς ή τον Διευθυντή, παρακαλώ. Κύριε Διευθυντά, ενδεχομένω. Όχι, δεν έχετε να πείτε κάτι. Πολύ ωραία. Απλώς να σα ευχαριστήσω και εγώ ως εκτελεστικός ε, διευθύντη τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Ελέγχου Ελίας, να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή Ελίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σχέδιο έκθεσης όσον αφορά την απαλλαγή για την εκτέλεση του προπολισμού του 2012. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να πετύχουμε τους στόχους της κοινή ε, αλληλευτικής πολιτικής. Χαίρομαι βεβαίως ε, για την αναγνώριση που μας παρέχεται. Πιστεύω ότι η έκθεση θα ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο το προσωπικό μας να συνεχίσει το σκληρό έργο. Μάλιστα θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την εκτέλεση, την ποιότητα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο πλαίσιο ακριβώ και της τήρησης των υποχρεώσεων μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσω ότι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι 20 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και συγχαρητήρια και πάλι. Σημείο 11. Απαλλαγή. Όσον αφορά τον γενικό προπολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκδώσουμε έκθεση όπως κάναμε και για το προηγούμενο θέμα. Ανατέθηκε το καθήκον στον πρόεδρο της Επιτροπής μας. Αντίστοιχα με τα περσινά βεβαίω. Έχουμε τις ενισχύες μας, έχουμε προτάσεις, είναι λίγο πολύ τα ίδια όπως είπαμε αυτά που είχαμε γράψει και πέρσι. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου δεν περιέχει επαρκείς λεπτομέρειες για τα ζητήματα της θάλασσας. Και συναφώς και της αλίας. Όπως ε, είπα και για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου Αλίας, ε, ο προπολογισμός έχει εκτελεστεί σε πολύ ψηλό ποσοστό, αν και δεν υπάρχουν γενικότερα στοιχεία. Πάντως, επαναλαμβάνω, η εκτέλεση, η υπορρόφηση είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα παρατήρησή μα είναι ότι μάλλον το ελεγκτικό συνέδριο ε, σημειώνει ένα δικαιολογητά υψηλό ποσοστό λαθών σε σύγκριση με την περισμένη χρονιά. Αν και βέβαια ε, αυτό πρέπει να συνδυαστεί με το γεγονός ότι το ελληνικό συνέδριο άλλαξε την μέθοδο δειγματοληψίας. Δεν υπάρχει ξεχωριστός δείκτης ε, σφάλματος για την Ελία, οπότε δεν μπορούμε ε, να συνεργάζουμε συμπεράσματα. Ζητούμε όμως να υπάρχει ξεχωριστό δείκτη τα επόμενα χρόνια. Σημειώνουμε επίσης την επιφυλάξη της DG Mare. Ειδικά όσον αφορά ένα πρόγραμμα που χρονολογείται από το 2001. Αυτή την επιφύλαξη πρέπει να την δούμε. Καλή είναι η έλεγχη και τη θεωρήση, αλλά πρέπει τα θέματα κάποια στιγμή να κλείνουν. Για την προστασία βεβαίω των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν τομεί επίσης κοινή διαχείριση για διαφορέ πιστώσεις. Ας προσπαθήσει και η Γενική Διεύθυνση Μάρε να κάνει ό,τι χρειάζεται για να αρθούν και οι σχετικές επιφυλάξεις από τους ελεγκτές. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε επισημάνει. Κάθε επανάληψη είναι επί ετών και αφορά την εξωτερική διάσταση της θαλασσίας πολιτικής και της πολιτικής ελίας. Όπως και με τις προηγούμενες εκθέσεις, κατά κλειδί χορηγούμε απαλλαγή για την εκτέλεση του προπολογισμού του 2012. Θέλει κανεί το λόγο. Σχόλια παρακαλώ. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών. 20 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Πολύ ωραία. Θεωρώ η γνωμοδότηση εγκρίνεται και περιμένουμε τροπολογίες βεβαίω. Επόμενο σημείο παρουσίασε θεματικό τμήμα Β ενημερωτικού σημείωματο με τίτλο Συνεργασία Τρομέα τη Ελία με Ισλανδία και Νορβηγία. Δεν έχει έρθει ο μιλητή ο κ. Ρότζερ, οπότε α διακόψουμε για 10 λεπτά μέχρι να έρθει ο κ. Ρότζερ, ο μιλητή για το 12. Ή είναι εδώ. Ήρθε. Όχι, λοιπόν, διάλειμμα 10 λεπτών. Κρίμα δεν είναι εδώ, αλλά ούτω ή άλλω ε, Δεν έχουμε συγκεκριμένο ωράριο, αλλά αν και λέω στον κόσμο να έχετε πιο νωρί. Εν πάση περιπτώσει, 10 λεπτά διάλειμμα. δεν θα

Okay, ladies and gentlemen, can we... Κυρίες και κύριοι, μπορούμε παρακαλώ να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Έχουμε φτάσει στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης, που είναι παρουσίαση του Τμήματος Πολιτικής 5 και αφορά την ε, συνεργασία στον τομέα της αλίας με την Ισλανδία και την Ορβηγία. Την παρουσίαση θα την κάνει ο Dr. P. E. Rogers, που είναι σύμβουλος από την εταιρεία Erinshaw Economics Limited. Είναι λοιπόν χαρά μου που καλωσορίζω τον δόκτωρα Ρότζερς στην Επιτροπή Αλίας. Ε, χωρίς πολλά πολλά λοιπόν, σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με ακούτε όλοι η πρώτη μου ερώτηση. Ωραία. Το έγγραφο αυτό έχει να κάνει με την συνεργασία στον τομέα της αλληλείας ανάμεσα στην Ισλανδία και την Ορβηγία. Ο στόχος του εγγράφου ήταν να εξεταστεί η παρούσα κατάσταση στην Αλία. Έχουμε κάποια ε, μεταναστευτικά είδη και επικαλυπτόμενα είδη στον Βόρειο Ατλαντικό. Μιλάμε δηλαδή για αποθέματα που μετακινούνται ανάμεσα στις ε, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των παράκτιων κρατών. Και υπάρχουν και τα επικαλυπτόμενα είδη, τα οποία ζουν και από τις δύο πλευρές των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες δεν καλύπτουν όλες τις, όλα τα ύδατα του κόσμου, το οποίο σημαίνει ότι αυτά τα αποθέματα ε, μένουν και σε διεθνή ύδατα. Αλλά τα είδη για τα οποία μιλάμε τώρα, που είναι το προσφυγάκι, ο καπελάνος, το η Ρέγκα, το Σαβρίδι, το Σκουπρί και η Σαρδέλα έχουν ως χαρακτηριστικό ότι είναι πελαγικά είδη. Είναι είδη που μετακινούνται σε κοπάδια για να βρουν τροφή και να αναπαραχθούν. Το πεδίο της μελέτης αυτής ήταν κυρίως να εξετάσει την περιοχή ISIS 27 και ιδιαίτερα βόρεια του γεωγραφικού πλάτους 62. Βλέπετε ότι έχουμε ρωσικά ύδατα, ύδατα της Γρυλανδίας, στα δυτικά, νορβηγικά, γύρω από το νησί Γιάν Μάγεν και στην ε, νορβηγική ακτή, ε, ύδατα της Ισλανδίας, ε, των Φερών Νήσων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης διεθνή ύδατα. Η διεθνής περιοχή που μας ενδιαφέρει εδώ πέρα είναι αυτό το παράθυρο που βλέπετε στα βόρεια. Η παρουσίαση ακολουθεί την διαδομή με το έγγραφο που σας έχω υποβάλει. Πρώτα θα σας παρουσιάσω κάποια γενικά στοιχεία, κατόπιν θα αναφερθούμε στα γενικά ρυθμιστικά μέτρα της αλληλείας και θα εξετάσουμε δύο περιπτώσεις, ε, τη Ρέγκα και το Σκουμπρί. Θα εξετάσω κατόπιν τον αντίκτυπο τη μεταρρύθμισης τη κοινή αλληλευτική πολιτικής που θα τεθεί σε ισχύ τον επόμενο μήνα. Θα εξετάσουμε μετά τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας, ιδιαίτερα με την Ισλανδία και την Ορβηγία. Ε, συμπεριλαμβάνω όμω και τι Φερόε νήσους ω ξεχωριστή οντότητα στο έγγραφο αυτό. Πρόκειται για διοικητικό παράδειγμα της Δανίας. Έχει λοιπόν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ξεχωριστή οντότητα τις Φερόες νήσους. Κατόπιν θα εξετάσω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στις συζητήσεις ε, για την αποκατάσταση αυτών των αποθεμάτων και το τι συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε και τι θα πρέπει να γίνει. Πρόκειται για κάποια από τα πλησιότερα λευτικά πεδία του κόσμου το βάθος των υδάτων, ε, η διαθεσιμότητα ε, τροφίμων, ε, τροφής σημαίνει ότι έχουμε εδώ πολύ μεγάλα αποθέματα, αλλά τα πελαγικά είδη στα οποία αναφέρθηκα νωρίτερα, μένουν ή περνούν από διάφορες αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και Επίσης, μένουν ή μετακινούνται και σε διεθνή ύδατα. Βλέπουμε λοιπόν ότι περνούν από διάφορε ζώνε. Ε, οι αληθικοί στόλοι προέρχονται από τη Δανία, τι Φερόε, την Ισλανδία, Ιρλανδία, κάτω χώρε, ε, Νορβηγία, Ρωσική Ομοσπονδία και Σκοτία και σε λιγότερο βαθμό ε, προέρχονται από άλλε χώρε συμπεριλαμβανομένε τη Γρυλανδία. Έχουν προκύψει προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Το σύστημα Σύναψη συμφωνιών για τα τάκ και τις ποσοστώσεις για τους εθνικούς στόλου έχει καταρρεύσει. Το θέμα που τίθεται είναι γιατί. Είχαμε στην Ευρώπη μια τεράστια οικονομική κρίση μετά την ε, τραπεζική κρίση του 2008. Το πρόβλημα είναι οι οικονομικές πιέσεις συνέβαλαν στην κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. Η Ισλανδία και η Φερόες εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αλληλεία για το εισόδημά τους. Το ΑΕΠ τους εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αλληλεία. Ιδιαίτερα οι Ισλανδοί, προσπάθησαν να, να διαφοροποιήσουν την οικονομία τους με τον τραπεζικό τομέα. Θα θεωρούσε κανείς λοιπόν ότι οι οικονομικές πιέσεις αυτές μπορούν να συνέβαλαν στην κατάρρευση των συνομιλιών. Λόγω της πίεσης στους διαπραγματευτές να πετύχουν όλο και περισσότερα. Αλλά από ό,τι φαίνεται τελικά αυτό δεν ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βλέπετε τον συντελεστή ανάπτυξη. Η Ισλανδία συνέρχεται. Η ανεργία είναι αρκετά ψηλή, όχι όμως υψηλότερη στη Δυτική Ευρώπη, στην Ισλανδία. Δεν φαίνεται λοιπόν οι οικονομικές πιέσεις να συνέβαλαν στην κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, των συμφωνιών. Ποιες είναι λοιπόν οι συμφωνίες αυτές. Έχουμε την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ε, για τον νόμο της θάλασσας, ε, που σημαίνει ότι τα παράκτια κράτη είναι από κοινού υπεύθυνα για την ε, βιώσιμη διαχείριση των αλλιευμάτων. Και παράκτια κράτη είναι αυτά μέσω των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των οποίων περνούν τα αλλιεύματα. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί εφόσον συμφωνηθούν τάκ, και εφόσον εφαρμοστούν από τα σκάφη των παρακτήων κρατών. Η διαχείριση πραγματοποιείται σύμφωνα με την Συμφωνία του 1995 των Ηνωμένων Εθνών, η οποία δημιούργησε την ε, Επιτροπή Αλληλείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού. Τα κράτη που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των παρακτήων κρατών εξαρτάται από το απόθεμα. Η Επιτροπή λοιπόν του Βορειοανατολικού Ατλαντικού θέτει τα ΤΑΚ και κατόπιν επιτρέπει στα παράκτια κράτη να καταλήξουν σε συμφωνία ώστε να κατανεμηθούν οι εθνικές ποσοστώσεις. Όμως, όπως σας είπα, συμφωνία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, ιδιαίτερα για τη Ρέγκα και για το Σκουμπρί τα τελευταία χρόνια. Το σύστημα είναι κατακαιρματισμένο. Υπάρχουν κάποιες ποσοστώσεις που θεσπίζονται μονομερός σε εθνικό επίπεδο ή διμερός ανάμεσα σε κάποιες χώρες. Θεσπίζονται σε διάφορες χρονικές στιγμές και το σημαντικότερο είναι ότι οι ποσοστώσεις δεν αντικατοπτρίζουν τις επιστημονικές συμβουλές των βιολόγων της ISIS όσον αφορά τα ασφαλή επίπεδα εκμετάλλευσης. Η αλία σκουμπριού είναι ίσως η πιο σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα το σκουμπρί αποτελεί αντικείμενο με υψηλή ζήτηση από το κοινό. Εάν κοιτάξετε τη δεκαετία του 50, για παράδειγμα, η ζήτηση για το σκουπρί δεν ήταν πολύ υψηλή. Το 1974 η Ισλανδία είχε 5.000 τόνους, αλλά πέρα από αυτό δεν έχει αλλιεύσει πολύ σκουπρί. Μόνο γύρω στο 2008 έγινε σαφές ότι αυξανόταν η αλία σκουμπρίου γύρω από την Ισλανδία. Το 2009 η αλία σκουμπρίου ανερχόταν σε 100.000 τόνους. Είναι σημαντικό ο όγκος αυτός, το οποίο σημαίνει ότι είναι ένα από τα βασικά παράκτια κράτη όσον αφορά το σκουμπρί η Ισλανδία. Τελευταία φορά όμως που είχαμε επιτυχή θέσπιση ποσοστώσεων για το σκουμπρί ήταν το 2009. Έκτοτε οι Φερόες Νήσι και η Ισλανδία έχουν θεσπίσει μονομερό ποσοστώσει και οι Φερόες Νήσι έχουν καθορίσει το δικό τους τάκ για τη ρέγκα το 2013. Έχουμε λοιπόν κατακαιρματισμένο σύστημα, το οποίο είναι και υποξαφάνιση τελείως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νορβηγία κατέληξαν σε διμερή συμφωνία το 2010 για ένα δεκαετές ε, πρόγραμμα διαχείρισης του Σκουμπριού. Αυτό όμως ε, δεν το έχουν υιοθετήσει και η Φεροεσνήση και η Ισλανδία. Αυτή τη στιγμή αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ισλανδία και η Νορβηγία έχουν καταλήξει σε συμφωνία για, το για τα ΤΑΚ Σκουμπρίου για το 2014, όχι όμως και η Φεροεσνήση. Α κοιτάξουμε λοιπόν τις δύο περιπτώσεις. Έχουμε την ε, ρέγγα ιαρινής αναπαραγωγή ε, στην Νορβηγία. Βλέπετε στην αρχή του διαγράμματο αυτού ότι το απόθεμα αυτής της ρέγγα είχε καταρρεύσει. Αρχές ε, της δεκαετίας του 70 μάλιστα είχε καταστραφεί. Αυτό μάλλον οφείλεται στο Power Block, το οποίο διευκολύνει την ε, αλληλεία με γρηγρή ή πελαγικές στράτες. Ήταν ε, λοιπόν τρομακτικός ο αντίκτυπος στα αποθέματα ρέγγας... Ε, αλλά υπήρξε μορατόριουμ και βλέπετε ότι ως αποτέλεσμα αυτού άρχισε η αποκατάσταση των αποθεμάτων αυτών ε, στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Μέσα του 90, της δεκαετίας του 90 όμως αρχίσαμε να βλέπουμε αύξηση των εκφορτώσεων. Τα αποθέματα συνεχίζουν ε, να αποκαθίστανται λόγω των μέτρων διαχείρισης. Γύρω στο 2006 είχαμε την ε, ακμή, αλλά έκτοτε έχουμε πτώσει κατά 30%. Η μεσαία από τις τρεις γραμμές ε, είναι το απόθεμα αναπαραγωγής, όπου δεν βλέπουμε να υπάρχει πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά πάλι έχουμε μείωση ε, των εκφορτώσεων έχει αλλάξει το μοτίβο μετανάστευσης αυτής της ρέγγας. Βλέπουμε τέσσερις διαφορετικές διαδρομές μετανάστευσης. Η τελευταία φαίνεται στην οθόνη αυτή τη στιγμή. Οι αιτίες για τις ε, αλλαγές αυτές δεν είναι γνωστές. Από το 2003 και μετά το σκουμπρί έχει αυξηθεί σε επίπεδα που έχουμε να δούμε από τη δεκαετία του 70. Βλέπετε στην αρχή την... τις επιπτώσεις του power block. Κατόπιν είχαμε εισαγωγή νέων μέτρων διαχείρισης και βαθμία αποκατάσταση από το 2002 και μετά. Και Τώρα πια η ISIS μπορεί να προτείνει τάκ για το 2014 κατά 60% υψηλότερο από το τάκ για το 2013. Επίσης έχουν αλλάξει οι διαδρομές αποδημίας του σκουμπριού. Βλέπετε περίπου τις διαδρομές στην οθόνη. Όταν ήταν πολύ μικρό το απόθεμα, Οι διαδρομές αποδημίας ε, ήταν κατά μήκος της νορβηγικής ακτής κάποια στιγμή. Το γιατί τώρα πια τα ψάρια έχουν αρχίσει να μεταφέρονται προς την Ισλανδία και τα νησιά Γιάν Μέιεν δεν είναι γνωστό. Δύο λόγοι έχουν προταθεί. Αλλαγές ε, στη θερμοκρασία του νερού. Δεν είναι σαφές αν το σκούπρι προτιμάει τα πιο θερμά ύδατα ή αν το κρύλ που τρώνε είναι περισσότερο παρόν εκεί ή εάν απλά το αυξημένο μέγεθος του αποθέματος ε, κάνει τα ψάρια να πεινάνε και να ψάχνουν αλλού τροφή. Ωστόσο, οι μονομερείς και διμερείς ποσοστώσεις που έχουν καθοριστεί για το 2013 απειλούν να μειώσουν το απόθεμα του νορβηγικού, ε, της νορβηγικής ρέγκας αναπαραγωγής και μπορεί τελικά να έχουμε επίπεδα χαμηλότερα από το βιολογικά αποδεκτά ελάχιστο. Το σύνολο των ποσοστώσεων για το 2013 βρίσκεται πάνω από τα τάκ που προτείνει η ISIS και μπορούν κάλλιστα να οδηγήσουν σε μείωση του αποθέματος εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτό ισχύει και για το σκουμπρί. Ποιο είναι ο αντίκτυπο τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Η μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική έχει πέντε πτυχέ. Πρώτον, απαγόρευση των απορρίψεων. Δεύτερον, περιφερειοποίηση. Τρίτον, ε, κοινωνική διάσταση. Τέταρτον, μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Καθώς ε, και τα μεταβάσιμα δικαιώματα αλληλείας. Πρώτον, όσον αφορά την απαγόρευση απορρίψεων, η πελαγική αλληλεία γενικά είναι αρκετά καθαρή αλληλεία. Συνήθως έχουμε αλληλεία μόνο των ειδών στόχων αν και πότε πότε αλλιεύονται ψάρια μεγέθου μικρότερου από το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης. Ε, δεδομένης όμως τη φύση των μέτρων, μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά καθαρή η αλία. Πότε πότε έχουμε ανάμειξη των ε, κοπαδιών ρέγγας και σκουμπριού Οι προτινόμενες αλλαγές στην κοινή αλλιευτική πολιτική για απαγόρευση των απορρίψεων θα είναι συμβατή με το παρόν καθεστώς διαχείρισης. Η Νορβηγία ήδη εφαρμόζει απαγόρευση απορρίψεων. Δεν υπάρχει λοιπόν ιδιαίτερο πρόβλημα με αυτή την πτυχή της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Όσον αφορά την περιφερειοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι η πελαγική αλληλεία είναι διαφορετική από την, ε, βαθύβι... από την αλληλεία βαθύβιων ε, ειδών και βενθοπελαγικών. Έχει δημιουργήσει Περιφερειακή Πελαγική Συμβουλευτική Επιτροπή και πάλι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα όσον αφορά την περιφερειοποίηση. Όσον αφορά την κοινωνική διάσταση. Ακόμα και με την πιο βιώσιμη διαχείριση της αλληλείας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει κάποια μικρή μείωση της απασχόλησης. Αυτό σχετίζεται με τις τεχνικές εξελίξεις στον τομέα αυτών που επιτρέπουν στον τομέα αυτόν να απαιτεί περισσότερο κεφάλαιο αλλά λιγότερο εργατικό δυναμικό. Αυτό δεν είναι κάτι που περιορίζεται στην αλλήλεια. Συχνά χρησιμοποιώ το, δικαίω, το παράδειγμα ε, ενός χωραφιού 10 εκταρίων δίπλα στο σπίτι μου. Πριν 10 χρόνια, για την σοδιά την φετινή θα χρειαζόντουσαν πολλά πρόσωπα. Θα βοηθούσαν και οι γυναίκες και παιδιά. Ενώ πέρσι έγινε με έναν που οδηγούσε τη σχετική μηχανή για τη συγκομιδή του κρυθαριού και ε, δύο νέους που βοηθούσαν. Τρία άτομα σε σχέση με 50 πριν κάποια χρόνια. Αυτή λοιπόν είναι μια φυσική εξέλιξη. Τα τελευταία 50-100 χρόνια λοιπόν ε, θα δούμε μείωση της απασχόλησης στον τομέα της αλίας. Ωστόσο είναι δυνατόν με αποτελεσματική διαχείριση και αποκατάσταση των αλλιευμάτων, βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, να έχουμε αύξηση της απασχόλησης στον τομέα της αλίας. Και επίσης στη στεριά, στον τομέα επεξεργασίας, μεταποίησης, διότι θα υπάρχουν περισσότερα ψάρια η αποτελεσματική διαχείριση λοιπόν της αλληλείας θα πρέπει να βοηθήσει στην αναχέτηση της μείωσης στην απασχόληση. Τώρα, μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ο στόχος της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης είναι κάπως αβέβαιος στόχος και αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα με την αλία Ρέγκας και Σκουμπριού στον Βόρειο Ανατολικό Ατλαντικό. Δεν είναι καθόλου βέβαιο εάν τα παρόντα μεγάλα αποθέματα μπορούν να διατηρηθούν μόνιμα ή εάν αποτελούν αποτέλεσμα κάποιας ιδιαιτερότητας στο οικοσύστημα. Στη Βόρεια Θάλασσα, στις, στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, είχαμε μία αύξηση του γάδου. Τα επίπεδα ήταν πολύ ψηλότερα από ό,τι είναι φυσιολογικό για τα αποθέματα αυτά. Μία πιθανότητα που άκουσα είναι ότι ο λόγος γι' αυτό ήταν ότι τα αποθέματα ρέγκας ήταν πολύ μειωμένα και έτσι υπήρχε πολύ τροφή για τα αποθέματα γάδου. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν γιατί είναι τόσο μεγάλα τα αποθέματα σκουμπρίου αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε αν είναι μόνιμη αυτή η κατάσταση ή όχι. Αλλά έχουμε εδώ ένα δίλημα. Θα πούμε ότι δεν ξέρουμε και θέλουμε να διατηρήσουμε ψηλά τα αποθέματα για το μέλλον ή λέμε ότι αυτό είναι πιθανότατα προσωρινό φαινόμενο και θα ήταν κρίμα να χάσουμε την οικονομική αξία των αποθεμάτων αυτών βραχυπρόθεσμα, ελπίζοντας ότι θα έχουμε κάτι στο μέλλον. Μήπως απλά εξαφανιστούν τα ψάρια αυτά στο μέλλον χωρίς να τα έχουμε αλλιεύσει. Δεν το ξέρουμε, είναι σημαντικό δίλημα. Θα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε στους ε, στους ε, βιολόγους, να φροντίσουμε να υποφεληθούμε από το πλεονέκτημα αυτό όσο υπάρχει, χωρίς όμως ε, να προκαλέσουμε ζημιές για το μέλλον. Όσον αφορά τις μεταβάσιμες αλλιευτικές παραχωρήσεις. Πιστεύω ότι η μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής δεν θα οδηγήσει σε σύγκρουση στον τομέα αυτών. Αυτή τη στιγμή και οι πέντε πτυχές της ε, μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην συνεργασία στον τομέα της αλίας ε, με την Νορβηγία, την ε, Ισλανδία, ούτε και με τις Φερόες νήσους. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας. Εξετάζουμε φυσικά τα επικαλυπτόμενα είδη. Εάν κάποιο αποφασίσει να αλλιεύσει όσο γίνεται περισσότερο, αυτό σημαίνει ότι απομένουν λιγότερα για του υπολείπου και το βασικό πλεονέκτημα της συνεργασίας με την Ορβηγία, τις Φερόες Νήσους και την Ισλανδία είναι ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε το μεγαλύτερο κέρδος με προσαρμογή των ΤΑΚ στις συνθήκες. Έτσι μπορεί ο τομέας να προγραμματίσει τις επενδύσεις του και μπορεί να ξέρει ότι θα αποφέρουν λογικά οι επενδύσεις αυτές. Βέβαια, σε, σε οποιαδήποτε επιχείρηση ισχύουν κάποια πράγματα για τις επενδύσεις ε, και δεν είναι μικρότερος ο κίνδυνος στον τομέα της αλληλείας. Αλλά ταυτόχρονα οι διαχειριστές της αλληλείας πρέπει να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που προκύπτουν από τη διακύμανση στο μέγεθος των αποθεμάτων, που, μπορεί, που είναι κάτι που μπορεί να αποφευθεί. Κάποιες ε, παράκτηε κοινότητες εξαρτώνται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την αλληλεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γεγονό. Στην ε, βορειοανατολική Σκοτία ε, η οικονομία εξαρτάται κατά 35% από την αλληλεία. Στην Ισλανδία είναι ανάλογο το ποσοστό. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να βρούμε την σωστή ισορροπία και οι αλλαγές στην τεχνολογία που θα επηρεάσουν την απασχόληση θα πρέπει να μετριαστούν. Και δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τον καταναλωτή. Ο καταναλωτής θα ωφεληθεί από την μεγάλη προσφορά. Θα πρέπει να παρέχονται σωστές και αξιόπιστες πληροφορίες στους καταναλωτές και επίσης ο τομέας μεταποίησης θα πρέπει να γνωρίζει ότι ότι έχει αρκετό προϊόν για να μπορεί να συνεχίζει τις εργασίες του. Είχαμε το μορατόριουμ για τη Ρέγκα στη Βόρεια Θάλασσα τη δεκαετία του 80 και ένας οικονομολόγος από τις κάτω χώρες είπε ότι το μορατόριουμ ήταν μεγάλη επιτυχία και είχαμε ε, σημαντική αποκατάσταση του αποθέματος. Όταν τελικά εκφορτώθηκαν τα ψάρια, η υποδομή που είχε χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των ψαριών αυτών είχε εξαφανιστεί. Σε κάποιο βαθμό δεν υπήρχε πλήρης αποκατάσταση της αλίας ρέγγας που είχαν οι κάτω χώρες. Αυτό οφειλόταν στο μορατόριουμ διότι οι δεξιότητες το δίκτυο πολίσεων χάθηκαν. μεγάλη προσφορά ψαριών αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα κατά την εξαγωγή. Εάν λοιπόν μπορούμε να έχουμε τέτοια μεγάλη προσφορά, τόσο το καλύτερο. Νομίζω όμως ότι το πιο σημαντικό που μπορώ να πω είναι ότι η διαμάχη που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των παρακτιών κρατών έχει προκύψει λόγω της αλλαγής της συμπεριφοράς των μεταναστευτικών ε, και επικαλυπτούμενων ειδών. Τα μεγάλα αποθέματα που έχουμε αυτή τη στιγμή έχουν επίσης επηρεάσει την κατάσταση. Η αποδημία λοιπόν των ψαριών είναι σημαντικός παράγοντας. Πιστεύω ότι οι λύσεις για τα προβλήματα εξαρτώνται από τον καθορισμό ενός μακροπρόθεσμου συστήματος για την κατανομή των ΤΑΚ. Έχουμε ένα σύστημα για τα δυτικά ύδατα της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν... Δεν γίνονται κάθε χρόνο διαμάχες μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με το ποσοστό των αλλιευμάτων που δικαιούνται. Είναι πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις αυτές. Φανταστείτε πόσο δύσκολες θα ήταν αν θα έπρεπε να γίνονται διαπραγματεύσεις για κάθε ποσοστό, κάθε αλλιεύματος, για κάθε χώρα. Στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό προσπαθούμε να βρούμε ένα σύστημα ώστε τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν πάνω σε μια κλίδα κατανομής σχετικά σταθερή. Το μόνο που θα πρέπει να συμφωνείτε στην αρχή κάθε χρόνου θα πρέπει να είναι το ύψος του ΤΑΚ, το οποίο θα καθορίζεται με βάση τις επιστημονικές συμβουλές. Ένα τέτοιο τάκ θα καθορίζεται κάθε χρόνο και θα εφαρμόζεται κάποιοι κανόνες. Θα υπάρχει ένα μόνιμο, μια μόνιμη κλίδα μια τέτοια κλίδα κατανομής θα πρέπει να αναγνωρίζει όχι μόνο τις αλλαγές στο μέγεθος των αποθεμάτων, αλλά και τις αλλαγές στις ε, μεταναστευτικές διατρομές. Οι βιολόγοι θεωρούν ότι η αλλαγή στις μεταναστευτικέ συνήθειε των ψαριών μπορεί να οφείλεται στην αλλαγή του μεγέθους των αποθεμάτων. Θα μπορούσαμε λοιπόν να εξετάσουμε την περίπτωση η κατανομή να προσαρμόζεται στο μέγεθος των αποθεμάτων και στις μεταναστευτικές διαδρομές, να μην υπάρχει δηλαδή σταθερό ποσοστό. Δεν νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να εκπονηθεί ο τύπος για κάτι τέτοιο, απλά θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία στην αρχή. Αυτή θα ήταν δύσκολη διαπραγμάτευση, αλλά θα είχε κανείς διαπραγμάτευση μια και καλή. Θα μπορούσε να δοκιμαστεί το σύστημα για πέντε χρόνια και αν διαπιστωθεί ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί, να συνεχιστεί και στο μέλλον. Βασικό είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πάλι κάποια συμφωνία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε επί χρόνια να συνεχίσουμε να λιεύουμε σε επίπεδα που θα απειλήσουν τα αποθέματα. Το ΤΑΚ θα πρέπει να συμφωνείτε κάθε χρόνο. θα πρέπει να συμφωνηθεί μια κλίδα κατανομής ε, μεταξύ των παράκτιων κρατών. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Muchas gracias. Y ahora pasamos a un turno de preguntas. Ας α, ξεκινήσουμε με ένα γύρο συζήτησης. Κύριε son. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Δόκτρα Ρότζε για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εισήγηση. Όπως γνωρίζουμε, η Νορβηγία αποχώρησε από τις πρόσφατες ομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα το Συμβουλίο δεν μπορεί να ασχοληθεί μετά τις Βόρειες Θάλασσες λόγω απουσίας συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νορβηγίας. πρώτη φορά το Συμβουλίο Αλίας βρίσκεται περιορισμένο προς την εντολή του εν του νέου έτους. Θα δούμε πώς και πότε θα καταλήξουμε στη συμφωνία με την Νορβηγία ώστε να λύσουμε τα προβλήματα των ποσοστώσεων και των ΤΑΚ συμπεριλαμβανομένων των λευκών ψαριών. Ο λόγο για τον οποίο αποχώρησε η Νορβηγία είναι ο νέο υπουργό, νέο στα σχετικά καθήκοντα, ο οποίο συναντήθηκε με την κυρία Δαμανάκη και από ό,τι κατάλαβα συνέστησε ένα διψήφιο τάκ για το σκουμπρί και την Ισλανδία και σε αυτό θα αφορούσε και τις φεροές. Και η Νορβηγία απλώς είπε όχι. Έγινε μια σε περιορισμένη σύνθεση συζήτηση με την κυρία Δαμανάκη πρόσφατα. Δεν μας είπε τι νούμερο έδωσε στους ενδιαφερμένους. Ποιο είναι το διψήφιο αυτό νούμερο. Πάντως η Ισλανδία και οι Φερόες επέμεναν στο 15% η Με βάση τώρα την πρόταση για τι 889.000 τόνους, πρόταση πάνω από τι 540.000, θα μπορούσαμε, ίσως να μπορούσαμε να δώσουμε αυτό το διψήφιο ποσοστό. όμω το πρόβλημα είναι, και φαντάζομαι θα το γράψουμε και στην εκθεσή μας, ότι έχουμε μείωση των αποθεμάτων. Έχουμε αντιθέτω, πρόταση για αύξηση 64% του αλλιεύματος. Αν λοιπόν τα αποθέματα μειωθούν κατά το αντίστοιχο ποσοστό το 2015, θα βρεθούμε ξανά στα επίπεδα των 500.000 τόνων. Θα έχουμε δώσει λοιπόν το 30% του τάκ μας σε Ισλανδία και Φερόες. Θα έχουμε καταστρέψει λοιπόν τους Ιρλανδούς, τους Σκοτσέζους και Άλλου ελίοι σε άλλα κράτη-μέλη. Οι επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές για τους κοινοτικούς ελίους. Οπότε, ανησυχώ όταν λέτε στην εκθεσή σα ότι η Συμβουλή των Επιστημόνων ουσιαστικά είναι παροχημένη, χρονολογείται από δύο ετών. Δεν έχουμε στοιχεία για τα δύο τελευταία χρόνια. Ξαφνικά λοιπόν μας λέει κανεί 64.000 τόνους, 64% με συγχωρείτε για το 14. Με βάση όμω τα στοιχεία του 11, ε, νιώθω πραγματικά πολύ ανήσυχο. Λόγω τη συμπεριφορά τη Ισλανδία και των Φερών πέρσι, ορισμένοι εκτιμούν ότι τελικώ καταστρέψαμε ένα εκατομμύριο τόνων σκουμπριού, όταν η σύσταση ήταν για το μισό. Τα αποθέματα λοιπόν συνεχίζουν να μειώνεται και ξαφνικά βλέπω σύσταση για 900.000. Δηλαδή θα φτάσουμε να θανατώσουμε ένα εκατομμύριο τόνους, το οποίο σημαίνει ότι θα εξαφανίσουμε εντελώς το απόθεμα. Έτσι δεν πάμε πραγματικά πουθενά. Και το ίδιο έγινε με το προσφυγάκι. Δεν μπορείτε να, πείτε λοιπόν στους ε, τέρους μας ότι μπορείτε να συνεχίσετε να ψαρεύετε στα παλιά επίπεδα και ταυτόχρονα να περιορίζουμε τους δικούς μας. Θέλουμε μια ισότιμη λύση. Η λύση που προτείνεται κατά άλλα είναι λογική. Ετήσιο τάκ σε αρτήσει και των μεταναστευτικών ροών των ψαριών. Σε αρτήσει των πραγματικών αποθεμάτων. Αν η κατανομή γίνει με γνώμονα τη σταθερότητα των αποθεμάτων, τότε, όπως λέτε και εσείς, αυτό μπορεί να αποτελέσει ισότιμη λύση. Όμως η Ισλανδία και οι Φεροές δεν έχουν καμία όρεξη να διαπραγματευτούν επί αυτή τη βάση. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση η οποία δεν εμπνέει και πολύ αισιοδοξία. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να οριοθετήσουμε, τα προβλήματα αυτά ε, των βόρειων θαλασσών και αυτό ακριβώς κάνει αυτή η έκθεση. Αναφέρει μία λύση που ίσως ε, να είναι και εφαρμόσιμη. Πρέπει λοιπόν να δούμε ε, πώς θα έχουμε, πώς έχουμε την καλύτερη αλληλεία και τα καλύτερα αποθέματα και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τα διατηρήσουμε και να τα εκμεταλλευτούμε με βιώσιμο τρόπο, αηφόρο. Ε, υπάρχουν ε, τρόποι να παρακολουθήσουμε τις μετακινήσεις των ψαριών, την αποδημία τους, να δούμε ακριβώς πώς κινούνται, να είμαστε κι εμείς ευέλικτοι, ε, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε και να εκμεταλλευτούμε τις γνώσεις που έχουμε και τα χαρακτηριστικά των ψαριών αυτών. Οι Ισλανδοί λένε πως ε, ψαρεύουμε συνέχεια τον ε, μπακαλιάρο ε, και τώρα που άλλαξε πορεία, άλλαξε ε, ρότα, τι θα κάνουμε. Μα εγώ πιστεύω μόνο μέσω των διαπραγματεύσεων και της συζήτηση και εκμετάλλευση των γνώσεων μπορούμε να βρούμε λύση. Σας ευχαριστούμε κύριε Νίλσον και κυρία Λοβίν. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, εισήγηση που μας κάνατε. Πρόκειται για μια περίπλοκη και πραγματικά ε, συναρπαστική κατάσταση. Και όλοι μας, ε, όχι μόνο στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά παντού πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Να λάβουμε υπόψη της κλιματικές αλλαγές, την βιοχημία ε, στην ε, θάλασσα. Ε, είναι όλα αυτά τεράστια σημασία στα ψάρια, αλλάζουν πορεία, τα νούμερα, ε, τα στόκ, υπάρχουν ε, ε, είδη που, τα οποία είναι πολύ επιθετικά και ξαπλώνονται που δεν τα είχαμε παλιότερα. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση δηλαδή. Θα πρέπει ωστόσο να προστατεύσουμε τα, τα είδη τα οποία αλλιεύουμε και τρώμε, να συνεχίσουμε την αλληλεία με βιώσιμο τρόπο έτσι ώστε να είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε ένα σύνολο κανόνων. Οι ποσοστώσεις της ε, Ιρλανδίας είναι τεράστιες και αυτό δεν είναι απαραίτητο καλό. Και οι Φερόες νήσοι έχουν προσφύγει στο διεθνέ Δικαστήριο για τη Θάλασσα. διότι έχουν επιβληθεί κυρώσει εις βάρος των φερόνισων. Επειδή μονομερός έθεσαν την ποσόστοση για τη ρέγγα. Από ό,τι φαίνεται μπορεί η Φερόες Νήσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσουν να προσεγγίζουν ένα τον άλλον. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε τις κλίδες κατανομής που θα λαμβάνουν υπόψη τους πολλά διαφορετικά κριτήρια. Να μην σχετίζονται δηλαδή μόνο με τα ιστορικά δικαιώματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε κάποια αποθέματα τα οποία καλύπτουν πολλές διαφορετικές ε, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και έχουμε κάποιες κλίδες κατανομής που θεσπίστηκαν πριν 10, 20, 30 χρόνια, πριν πολύ καιρό δηλαδή. Δεν θα πρέπει να θεωρηθούν λοιπόν τόσο αυστηρές και άκαμπτες οι ποσοστώσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμοστούν πάνω από ένα κριτήρια. Είναι σημαντικά τα ιστορικά δικαιώματα αλληλείας, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και άλλους παράγοντες, όπως πρότεινε και ο Φίλιπ Ρότζερς. Το μέγεθος του αποθέματος μπορεί να είναι ένας τέτοιος παράγοντας. Εάν λοιπόν το σκουμπρί και η Ρέγκα, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη μετακινείται βόρεια ή εάν έχει αυξηθεί, δεν παίζει ρόλο, αλλά καλό θα είναι να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Είναι σημαντικό όλες οι χώρες ε, του Βορείου Ατλαντικού να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να αλλιεύουμε με τρόπο βιώσιμο και να είμαστε ανοιχτοί ώστε να μπορέσουμε να εκπονήσουμε ένα σύστημα δίκαιο για όλους. Πρέπει να μοιραστούμε τον πλανήτη αυτόν και αυτή είναι η θέση μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Στήλε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ για την εισήγηση. Θα σήμερα γιατί είμαι μέλος της αντιπροσωπείας για την Ορφηγία και την Ισλανδία. Δεν είναι εδώ επικεφαλής μας, αλλά εν πάση περιπτώσει μας ενδιαφέρει το θέμα και ως αντιπροσωπεία και ως επιτροπή. Όπως είπε και ο μιλητής, πρέπει να βρεθεί ισορροπία. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες. Είπε και ο κύριος Στίβενσον όμως, είναι κρίμα που τα στοιχεία που έχουμε είναι παροχημένα. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ εκπρόσωπο του Συμβουλίου τη Κομισιόν. Πάντως, όσον αφορά τι συνομιλίες με τι φεροέ. Ε, και το γιατί έφυγαν, απεχώρησαν οι Νορβηγοί από τι συνομιλίε. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Οι Ισλανδοί και οι Νορβηγοί τέλη Μαρτίου θα είναι στην Νορβηγία και θα προσπαθήσουν να πάνε στι Φερόε. Στο τέλο εκείνη τη εβδομάδα πιστεύω ότι είναι σημαντικό όταν επισκεφτούμε τι Φερόε τέλη Μαρτίου, νομίζω 25-26 Μαρτίου. Πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εν μεταξύ εμεί τουλάχιστον καταλήξει και να στείλουμε το μήνυμα στι Φεροέ. Δεν ξέρω τι με όσα συμβαίνουν, αν με όσα συμβαίνουν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε λύση, δύσκολο, αλλά το συμφέρον είναι κοινό εν τέλει. Είναι κοινή διαχείριση των αποθεμάτων. Θα ήθελα λοιπόν και ξέρω ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι πρέπει η προσωπία να στείλουμε το σωστό μήνυμα στην Ορβηγία και Ισλανδία και Φεροές Χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Αυτό θέλω να πω με την ευκαιρία. Ε, απουσίασα 10 χρόνια από την Επιτροπή Ελίας και χαίρομαι που επιστρέφω και βλέπω και οικία πρόσωπα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρία Στυβίτς. Καλώς ήρθατε. Είναι η πρώτη φορά, αλλά όχι και η τελευταία, ελπίζω. Ο κύριος ε, Ρότζερ ο θα απαντήσει όλα. Ελπίζω. Παρακαλώ, κύριε Ρότζες. Πρόεδρε. παροχημένα στοιχεία. Δεν ευθύνη των επιστημόνων. Κάνουν ό,τι μπορούν. Γιατί κάποιο πρέπει να συλλέξει πρώτα τα στοιχεία. Για να τα αναλύσουν οι επιστημονέ. Λοιπόν, ξαν... ξαναλέω, δεν φτάνουν οι επιστημονέ. για το παροχημένο των στοιχείων. Τα στοιχεία κάποιο τα συλλέγει. Και οριστικοποιούνται στο τέλος της χρονιάς, μετά τα επεξεργαζόμαστε ένα χρόνο και ετοιμαζόμαστε μετά για την επόμενη χρονιά, κάνουμε τις προβλέψεις μας και ούτω καθεξής. Όπως γίνεται και με τα οικονομικά μοντέλα. Τι γίνεται στην οικονομία γίνεται και στα βιολογικά δεδομένα. Εκεί που ξέρετε, κατά τα άλλα που υπάρχει σταθερότητα δεν έχουμε πρόβλημα. Η αστάθεια είναι το πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε λίγο πιο πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το απόθεμα και τις συστάσεις όσον αφορά τα μέγιστα λιεύματα, τα τάκ. Ένα ακόμη πιο σημαντικό πρόβλημα πάντως όσον αφορά τα, τις συστάσεις της Επιτροπής είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία εκφορτώσεων για Ισλανδία, και Για μερικά χρόνια μάλιστα, όχι μόνο δύο. για αίσες θεωρεί οι ποσότητες που δηλώνουν είναι και οι αλληλευθύσεις ποσότητες. Αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας και δεν ευθύνει των επιστημόνων να πούνε ή όχι. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε αν έτσι όντως έχουν τα πράγματα. Δεν ξέρουμε αν οι ποσοστώσει όντω ελιεύονται ή υποαλλιεύονται ή υπεραλλιεύονται. Τώρα οι Ισλανδοί και οι Φερόε προσπαθούν να αποστρέψουν το μέλλον τους και δηλώνουν ποσοστώσει ακόμα και δεν τι έχουν αλλιεύσει. Καλύτερα πόσα λοιπόν. Πρόκειται για μια μαύρη τρύπα αν θέλετε. Είμαστε στο σκοτάδι και αυτή είναι η δυσκολία εν προκειμένου. Και αυτό λέω ότι έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία να καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία για να ξεπεράσουμε αυτόν τον σκόπελο. Χρειαζόμαστε στοιχεία. Χρειαζόμαστε ενημερωμένα στοιχεία. Πρέπει να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι γίνεται. Κατάλα. Κύριε Πρόεδρε, μακάρι οι Ισλανδοί και οι Νορβηγοί να μας στείλουν κάποια ενημέρωση, ένα αντίγραφο από τα στοιχεία τους. Ε, δεν θέλω να σας δυσκολέψω, είναι πολιτικό το θέμα, αλλά χθε το Συμβούλιο Υπουργών Αλίας Φερόες είπαν ότι θα διαπραγματευθούν για το σκουμπρί εάν άρει για την ρέγγα, τον περιορισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συμφωνούσατε με κάτι τέτοιο. Ε, συγγνώμη που σας τριμώχνω, είναι, ξέρω ότι είναι πολιτικό το θέμα. Πώς το βλέπετε όμως. Δεν ξέρω πώς θα κόστε, τι θα κόστη να συμφωνήσουμε. Είναι οικονομικό το θέμα. Αν ήξερα, αν είχα τα οικονομικά στοιχεία θα απαντούσα. Τέλος πάντων, είναι κάτι που δεν θα το λύσουμε εδώ, πόσο θα κοστίσει. Άλλη ερώτηση. Όχι. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Ρότζερς. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για την εισηγήσή σας. Και περνούμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Διάφορα. Υπάρχει κάτι στα διάφορα. Όχι. Πολύ ωραία. Το επόμενο, 14, ανακοινώσει του Πρόεδρου σχετικά με τι αποφάσει που έλαβαν οι συντονιστέ. Το μοιράσαμε, το έχετε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε, α, κύριε Φράγα. Κύριε Φράγα. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τι αποφάσει που λήφθησαν, αλλά να μην ξεχνούμε στο 2-1 για την παρανομή αρχελία και τα κριτήρια για τις χώρες που είναι στη μαύρη λίστα, που, τις μη συνεργαζόμενες χώρες εννοώ, να μην ξεχνούμε, επαναλαμβάνω, την πρόταση της Κομισιόν. Να έρθει εδώ και να μας πει για αυτά τα περίφημα κριτήρια και το πώς εφαρμόζονται. Και κάτι σχετικό. Θα ήθελα να προχωρήσουμε να οργανώσουμε αυτή την ακρόαση με την Επίτροπο, γιατί είχε πει ότι θα έρθει να μας μιλήσει. Πρόεδρος, βεβαίως, το προσθέτουμε στις ε, προτάσεις. Να το πούμε στην Κομισιόν ότι θέλουμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα, να έχουμε εδώ την Επίτροπο για να ακούσουμε ότι θέλουμε να ακούσουμε από την καθήλυνα αρμόδια. Πολύ ωραία, το καταγράφω ως πρόταση και αυτό, εξαιρετικά. Α, 22 Ιανουαρίου, 22 και 23 Ιανουαρίου θα ξανασυνδριάσουμε. Δεν έχω κάτι άλλο. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα σε όλους και καλή χρονιά. Ευχαριστώ που ήρθατε. Θα τα πούμε σε ένα μήνα γεμάτη ενέργεια και ανανεμένη. Γεια σας.